Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είναι ντροπή αυτά που γίνονται. Εγκαταλείψαμε αυτούς που αγωνίστηκαν το Ισλαμικό κράτος. Στην πρώτη γραμμή είναι πραγματική ντροπή. 300.000 μετατοπιστέντες. 70.000 παιδιά, όπω λέει η UNICEF, που υφίστανται τα πάνδυνα. Η παράνομη εισβολή τη Τουρκία που είναι κατά του διεθνού. δικαίου. Το ότι το δέχεται ο Τραμπ θα έπρεπε να το περιμένουμε. Το ότι δεν έγινε τίποτα από πλευρά Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πραγματικά ντροπή. Δεν πρέπει μόνο να καταδικάσουμε την στρατιωτική επέμβαση της Τουρκίας. Πρέπει να απαιτήσουμε να αποσυρθούν τα στρατεύματα και να ασκήσουν το ρόλο του στα Ηνωμένα Έθνη, να ξεκινήσει ο, ο πολυμερή διάλογο για την περιοχή, το πλαίσιο τη Γενέβη, να, γίνει ε, να γίνει σεβαστή η Συμφωνία 1325 του Συμβουλίου Ασφαλεία. Πρέπει να υπάρξει αποστολή των Ηνωμένων Εθνών στην περιοχή. Επίση, πρέπει να αναλάβουμε και τι δικέ μα ευθύνε. Δεν είναι δυνατόν να ανεχθούμε ο Ερντοάν να ε, επιστρέψει σε αυτή την περιοχή τους πρόσφυγες. Πρέπει να ανοίξουμε δυνατότητες ε, μετεκατάσταση ε, για τους πρόσφυγες αυτούς. Δεν κάνουμε τίποτα εδώ και τόσο καιρό. Τι γίνεται με τους εξοπλισμούς. Δεν πήρα μια απόφαση που να πηγαίνει πέρα από τις νέες άδειε πώληση όπλων. Πρέπει επίσης να επιχειρήσουμε να σταματήσει η εξαγωγή όπλων για τα οποία έχει ήδη δοθεί η άδεια. Κοιτάξτε, στη Συρία αποτύχαμε. Θα πρέπει να σταματήσουμε να είμαστε θεατέ, να αναλάβουμε τι ευθύνε μα. Γιατί η ανθρωπιστική κρίση, κρίση είναι επίση ευθύνη μα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Βιλίμ ένα Ευχαριστώ, κυρίε και κύριοι. Για άλλη μια φορά συζητάμε για την Τουρκία. Για άλλη μια φορά συζητάμε για τον Ερντοάν. Ε, όχι λόγω επιθέσεων ε, κατά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της εσωτερικής κατάστασης στην Τουρκία. Όχι, αυτή τη στιγμή έχουμε έναν επιθετικό πόλεμο στη Βόρεια Συρία που αποσταθεροποιεί την ευρύτερη περιοχή. Και ποιο χάνει για άλλη μια φορά, κυρίω οι Κούρδοι που τα τελευταία χρόνια ποτέ δεν είχαν την αναγκαία στήριξη τη διεθνού κοινότητα. Είναι ο μεγαλύτερος λαός ε, του πλανήτη χωρίς κράτος θα πρέπει επιτέλους να υπάρξουν οι αναγκαίες επιπτώσεις. Και από ό,τι μαθαίνουμε, κάποιοι μαχητές του Ισλαμικού κράτους επιστρέφουν στην Ευρώπη για τα απελευθερώθηκαν. Πρέπει οπωσδήποτε να, να σταματήσει το καθεστώς υποψήφιας χώρας και να μην δίνουμε βοήθεια στην Τουρκία. Και να σκεφτούμε τι κυρώσεις μπορούμε να επιβάλλουμε. Και εμπάργο όπλων οπωσδήποτε να επιβληθεί. Η κατάσταση όπως είναι τώρα είναι απαράδεκτη. Σας καλώ, σας έγκαλώ να μην βάλουμε για άλλη μια φορά το κεφάλι στην άμμο. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Βάιμερς, ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η επέμβαση της Τουρκίας στην Βόρεια Συρία αποδεικνύει τη διαφορά μεταξύ ελέγχου των συνόρων και εξωτερικής πολιτικής. Λόγω της αφέλειας της δύση. χορηγήσαμε τον έλεγχο των εξωτερικών μας συνόρων στην Τουρκία. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα λόγω της μόνιμης απειλής ότι η Τουρκία μπορεί να ανοίξει τη στρόφιγγα στους πρόσφυγες. Η Τουρκία μας έχει στο χέρι. Η κυρία Μογκερίνη το είπε. Η Τουρκία έχει αποσταθεροποιήσει την περιοχή. Έχει ε, δημιουργήσει πολλά θύματα μεταξύ των αμάχων. Έχει αυξήσει τον κίνδυνο τρομοκρατίας. Έχει θίξει τη συμμαχία κατά του Ισλαμικού κράτους. Την έχει αποδυναμώσει. Δεν είναι δυνατόν να δεχόμαστε αυτή την κατάσταση. Η Τουρκία δεν είναι δημοκρατικό κράτος. Δεν μπορούμε να προστατεύσουμε ούτε καν τον πληθυσμό μας. Ευχαριστώ. Ο κ. τα γεγονότα αποδεικνύουν ότι υπάρχει μια καθαρή συμφωνία μεταξύ Τραμπ και Πούτιν με βασικό παίκτη τον κύριο Ερντογάν. Μοιάζει σαν τη διαφήμιση γνωστή εταιρεία ουίσκι εδώ τη Δύση. Ο ένα φεύγει, ο άλλο έρχεται. Η χθεσινή συμφωνία του κύριου Ερντογάν με τον κύριο Πούτιν αποδεικνύει το λόγο του αληθέ. Η Ένωση παίζει για άλλη μια φορά το ρόλο της συμμετοχικής αποχής με το αζημίωτο φυσικά για κάποιες χώρες της. απαντώντας σε ερώτηση γερμανικής αριστεράς η γερμανική κυβέρνηση απάντησε ότι μέχρι το εμπάργκο μέχρι προχθές δηλαδή είχαν πουληθεί στην τουρκία 250 δισεκατομμύρια ευρώ από στρατιωτικά για όπλα δηλαδή μέχρι το πρώτο οκτάμινο του 19. Από αυτό το μακελιό φαίνεται ότι όλοι κερδίζουν. Εδραιώνοντας τον κύριο Ερντογάν κυρίαρχο παίκτη στο Λεβάντε όμω υπάρχουν κάποια ερωτηματικά που θέλουμε να θέσουμε ποιο θα εγγυηθεί το ένα εκατομμύριο ψυχέ κούρδων στην περιοχή η ένωση; τι θα πούμε για το νέο κύμα προσφυγιάς που θα πάρει το δρόμο προ την ευρώπη και τα ελληνικά νησιά; η ένωση; θα στείλουμε τη συμπόνια μα, θα κάνουμε μια νέα συμφωνία Ευρωπαϊκή Ένωση Τουρκία ή θα βλέπουμε τον κύριο, ορμπαν να κλείνει τα σύνορά του. η πολιτική πλειοψηφία τη Ένωση κάνει καθημερινά την ένωση όλο και πιο αναξιόπιστη στο διεθνέ παιχνίδι. Ευχαριστώ κύριος Τέναντ ε, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αναρωτιέμαι τι στο καλό θεωρεί η Τουρκία ότι κάνει με αυτή την στρατιωτική επίθεση στην βορειοανατολική ε, Συρία. Δεν έχουν καμιά ανθρωπιά. Δεν αναγνωρίζουν πώς έχει υποφέρει αυτό το έθνος από τον Άισις, από τους βομβαρδισμούς. Εδώ καθόμαστε και μιλάμε για την Τουρκία που παραμένει υποψήφια στα χαρτιά για ε, προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ε, ε, πραγματικά ε, ακούμε όλο καλά ε, λόγια για τον Ερντογάν και το καθεστώς του, ενώ στην πραγματικότητα αυτά που κάνει δεν συνάδουν με τη σύγχρονη δημοκρατία. Αυτοί λοιπόν που κάνουν τα στραβά μάτια δεν μπορούν να συνεχίσουν. Πρέπει να κοιτάμε στον καθρέφτη και να βλέπουμε τι έχουμε αφήσει να γίνει. Και πραγματικά θα, δεν θα αντισταθώ στον πειρασμό να σας πω, σας το έλεγα. Μία τόσο μακροχρόνια σύγκρουση όπως τη Συρία δεν χρειάζεται νέες παρεμβάσεις ε, μονομερείς. Η Τουρκία σημαίνει δεινά, σημαίνει θάνατη, μετατόπιση μεγάλων μημάτων του πληθυσμού και μπορεί να βοηθήσει και το Ισλαμικό κράτος διότι θα βοηθήσει να δραπετεύσουν διάφοροι μαχητές και θα επιτρέψει και μεγαλύτερη παρουσία της Ρωσίας στην περιοχή που γίνεται επιδιαιτητής της κατάστασης πολύ περισσότερο μετά τη χθεσινή συμφωνία στο Σότσι η έξοδος της, ε, των Ηνωμένων Πολιτειών από τη Συρία και η απουσία της Ένωσης δημιούργησαν κενό που καλύπτουν η Ρωσία, η Τουρκία και το Ιράν. Και όλα αυτά θα έχουν σοβαρές επιπτώσεις. Η Ρωσία παίζει λοιπόν αυτό τον ρόλο, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αυξήσει το ρόλο της. Δεν μπορούμε απλώς να δίνουμε ανθρωπιστική βοήθεια και να βοηθάμε την ανοικοδόμηση. Η Ένωση πρέπει να προβλέπει. Χρειαζόμαστε μια πολιτική εξωτερικών και άμυνας πολύ πιο ενεργή τα, οι δυνατότητες διεθνούς διακυβέρνησης όπως ε, το Συμβούλιο Ασφαλείας δεν παίζουν τον ρόλο τους ενώ η Ουάσιγκτον επιστρέφει στον απομονωτισμό. Πρέπει να είμαστε πιο φιλόδοξοι. Στην περίπτωση της Συρίας δυστυχώς αποδείξαμε την ανεπάρκειά μας. Ευχαριστώ πολύ. Ένα λεπτό η κυρία Νησιέρα. Κυρία Πρόεδρε, πραγματικά ντρέπομαι από την ευκολία που η, Ευρω... διεθνής ε, ε, ε, κοινότητα δείχνει να μιλάει για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στο σχέδιο του ψηφίσματος μιλάμε για ζώνες κατάπευσης του πυρός στη Ράζοβα και γενικά μιλάμε για μια ειρηνευτική αποστολή. Όμως ε, αυτά είναι λόγια που δεν αρκούν. Ε, θα πρέπει να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Ε, είναι μια εισβολή και πρόθεση είναι η κατοχή. Δεν είναι απλώς παρέμβαση και ε, ήρθα σε επαφή με ανθρώπους όπως ο Μοχάμετ 12 ε, χρονών ε, που έχουν υπάρξει θύματα αυτής της κατάστασης. Το μόνο έγκλημα του Μοχάμετ είναι ότι γεννήθηκε Κούρδος σε μια περιοχή που ελέγχει ο Ενδογάν και η Τουρκία. Και πραγματικά πριν από 50 χρόνια υπήρξε εισβολή στη Βόρεια Κύπρο ε, και πριν από δύο εβδομάδες ε, βλέπουμε ακριβώς ε, τον Ερδογάν να μπαίνει στη Συρία. Δεν πρέπει να καθόμαστε σιωπηροί κάθε φορά που αυτό συμβαίνει. Ο κύριος Αουστροβίτσιος για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Η χρήση της στρατιωτικής βίας δεν είναι σωστή προσέγγιση για να λύσουμε τις προκλήσεις για να λύσει η Τουρκία τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει στα νοτιοανατολικά της σύνορα αντίθετα προκαλεί νέες επιπλοκές επιτιθέμενη κατά των κουρδικών ε, δυνάμεων, η Τουρκία προκαλεί δεινά στους Κούρδους, του Σύριους και του δικούς της πολίτες. Πέρα από τις ε, απώλειες αμάχων, οι παλιές πληγές των πληθυσμών ξανανοίγουν. Η λυπηρή αποχώρηση των ΗΠΑ, η απόλυτα μη αναγκαία τουρκική στρατιωτική παρέμβαση και η καταστροφική ρωσική στρατιωτική και πολιτική παρουσία των Ρώσων στη Συρία δημιούργησαν μια αλλαγή στην γεωστρατηγική ισορροπία που δεν μπορεί να είναι βιώσιμη. Η Ένωση πρέπει να παίξει ενεργό ρόλο για να ασφαλίσει ότι η Τουρκία θα λογοδοτήσει και παρά να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να συνεχίσουμε τον ζωτικό διάλογο αλλά με επικρίσεις κατά της Τουρκίας. Οι Κούρδοι της Συρίας πρέπει να βρεθεί τρόπος να σταματήσουν τα μακροχρόνια δεινά Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. 1,5 λεπτών. Ο κύριος Αλφονσί. Κυρία Πρόεδρε, η εισβολή της Τουρκίας στην περιοχή της Ροτζάβα πραγματικά θέτει πολύ σημαντικά ερωτήματα για το μέλλον της Ευρώπης καταρχάς. Σταθερότητα όσον αφορά την περιοχή αυτή. Οι Κούρδοι δείξανε τεράστιο θάρρος μέχρι την νίκη κατά του Νταέσ, μολονότι η Τουρκία έδειξε και δείχνει ακόμα διτή διπλή στάση. Αυτή τη στιγμή λέει ότι στρέφεται κατά των Κούρδων λόγω της τρομοκρατίας, αλλά ουσιαστικά προωθεί αυτή τη στιγμή τρομοκρατία. Δικαιώματα των ανθρώπων, δικαιώματα των γυναικών. Το Κουρδιστάν αυτή τη στιγμή προτείνει ένα καινούριο μοντέλο απέναντι σε όλες τις μουσουλμανικές χώρες περιοχής. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ασφάλεια της Ευρώπης σε έναν κόσμο που γίνεται όλο και πιο επικίνδυνος και που χρειαζόμαστε όλο και περισσότερους συμμάχους. Πώς θα καταφέρουμε να εξασφαλίσουμε στο μέλλον συμμάχους αν δεν προστατεύουμε τους σημερινούς μας συμμάχους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να λάβει δράση από μόνη της επιβάλλοντας αποτελεσματικές και ισχυρές διπλωματικές και οικονομικές κυρώσεις. Το εμπόριο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τουρκίας είναι πάρα πολύ σημαντικό, πιο σημαντικό και από το εμπόριο που έχουμε με τις ΗΠΑ. Θα πρέπει λοιπόν ήδη από σήμερα να καταφέρουμε να επιβάλλουμε αποτρεπτικές κυρώσει κατά της δικτατορία του Ρετσέπ Ταγί Περντογάν. σα. ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Μάντισον τώρα έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, συμφωνώ με τους προλαλήσαντες οι οποίοι είπαν ότι η δράση της Τουρκίας στη βορειοανατολική Συρία είναι απαράδεκτη. Ωστόσο και οι κυρώσεις αυτή τη στιγμή τίθενται να αμφιβόλω. Σαφώς θα πρέπει να αναλάβουμε δράση, αλλά ποια μέτρα ακριβώς, ποια αντίμετρα εμεί μπορούμε να υιοθετήσουμε απέναντι στην Τουρκία. Η αριστερά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μα λέει ότι θα πρέπει να προωθήσουμε οικονομικέ κυρώσει. Συμφωνώ με αυτό. Από την άλλη, όμω, θα πρέπει να δούμε και το εξή. Η Τουρκία τα τελευταία χρόνια εκβιάζει την Ευρωπαϊκή Ένωση λέγοντα ότι αν δεν δώσουμε την απαραίτητη κοινοτική χρηματοδότηση προ αυτού, θα ανοίξουν τι πύλε και θα κατακλειστούμε με πρόσφυγε. Μα ήδη 6 δισεκατομμύρια ευρώ έχουμε δώσει τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Για ποιο λόγο γίνεται αυτό για να μας εκβιάζει εκ νέου τώρα η Τουρκία. Είτε μας αρέσει είτε όχι, οι Ηνωμένε Πολιτείε διαδραματίζουν ένα σημαντικότατο ρόλο και συμβάλλουν τελικά στη σταθερότητα της περιοχής. Αυτή τη στιγμή αποσύροντας σε μερικοί τα στρατεύματά της, αφήνει ένα πολύ μεγάλο περιθώριο δράσης πια στη Ρωσία και την Τουρκία. Ελπίζω να καταφέρουμε να επέμβουμε κι εμείς για να βελτιωθεί η κατάσταση. Ο κύριος Ρούισεν τώρα έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τα όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στη Βορειοανατολική Συρία είναι πραγματικά απαράδεκτα. Η ειρηνική συμφιλίωση μεταξύ χριστιανών Κούρδων σε ένα καθεστώς δημοκρατικής αυτοδιάθεσης έχει καταστραφεί πλέον εξαιτίας της ε, στρατικής αυτής επέμβασης της ε, Τουρκίας στη Βορειοανατολική Συρία με το με την ονομασία, την κωδική ονομασία πηγή ειρήνης που θυμίζει λίγο φράση από βιβλίο του Orwell. Νομίζω λοιπόν ότι ε, θα πρέπει να συντοπίσουμε ότι υπάρχουν και πάρα πολλοί μαχητές του ISIS αυτή τη στιγμή που είναι ελεύθεροι. Νομίζω ότι οδηγούμαστε σε ένα νέο καθεστώς αστάθειας. Πού είναι η Ευρώπη, μάλλον που ήταν η Ευρώπη, μπορώ να πω και λίγο νωρίτερα φέτο, όταν ε, οι Ηνωμένε Πολιτείε. Ε, ζήτησαν στρατιωτική υποστήριξη για τις Συριακές δυνάμεις και πάρα πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η μία μετά την άλλη, αρνήθηκαν να παράσχουν αυτή τη στρατιωτική υποστήριξη. Σίγουρα έχει υπερβεί τα αποδεκτά αυτή τη στιγμή η Τουρκία και προφανώς εμείς θα πρέπει να αντιδράσουμε στη στάση αυτή, αντί να δείχνουμε την πολύ ήπια αντίδραση, την πολύ αδύναμη αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Ας σταματήσουμε πλέον να αντιμετωπίζουμε την Τουρκία σαν ένα πιθανό μελλοντικό μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πραγματικά εμείς θα λυγίσουμε μπροστά στο στρατηγικό όραμα του Ερντογάν. Πριν από ε, μία εβδομάδα ο Ευρωπαίος ε, Επίτροπος για την ε, Μετανάστευση συναντήθηκε με τους Τούρκους και είπε ότι είναι τέρος κλειδί για τη μετανάστευση και είπε ότι εξακολουθεί να ισχύει η ξεδιάτροπη συμφωνία Ένωσης Τουρκίας. Αυτές οι δηλώσεις γίνονταν ενώ ο τουρκικός στρατός εισέβαλε στην Ροζάβα. Φαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση όχι μόνο κάνει τα στραβά μάτια, αλλά νομοποιεί τον πόλεμο του Ερντοάν κατά του κουρδικού λαού, που ε, στην ουσία είναι συνοροφυλακή, συνοροφυλακή της Ευρώπης Φρούριο. Πρέπει να καταδικάσουμε την εισβολή και την εθνοκάθαρση κατά των Κούρδων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να είναι συνένοχος ε, σε αυτά τα εγκλήματα. Οι συμφωνίες με την Τουρκία πρέπει να παγώσουν. Πρέπει να αξιοποιήσουμε όλες τις πιέσεις των λαών, των θεσμών, ό,τι χρειάζεται για να σταματήσει αυτός ο πόλεμος. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος ε, Ζόνεμπορν, ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, όταν με ρωτάνε τι δουλειά κάνω. Τους λέω ότι μόλι βγήκα από τη φυλακή και ψάχνω να βρω τι πρέπει να κάνω. Αυτά που έχουν να κάνουν με την Ένωση λοιπόν είναι πολύ δυσάρεστα. Δεν θέλω να τον πω. Διότι ο παλαβός του Βοσπόρου κάνει πόλεμο, σκοτώνει αμάχους με γερμανικά όπλα, ενώ το ΝΑΤΟ, η Ένωση και η Γερμανία τον βοηθάνε. Με το δικτάτορα πρέπει να μιλήσουμε γλώσσα που να την καταλαβαίνει. Και γι' αυτό λέω Εάν ο Ερντοάν μας απειλεί με 3 εκατομμύρια πρόσφυγες, τότε να τον απειλήσουμε κι εμείς με 3 εκατομμύρια Τούρκους από το Κρόιτσμπεργκ, να τα στείλουμε πίσω. Και αν δεν φτάνουν αυτά, θα στείλουμε από πίσω τους και 3 εκατομμύρια Γερμανούς συνταξιούχους. Έτσι, πρώτα απ' όλα, θα μειωθούν οι τιμές των ακινήτων στη Γερμανία και θα μειωθούν και οι ψηφοφόροι του Τσέντεου στη Γερμανία. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριο Λέναρ, Ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Πολλά υπόθηκαν για τη σύγκρουση στη Συρία και τη γεωπολιτική της διάσταση. Αλλά δεν είναι μόνο γεωπολιτικό θέμα. Είναι και θέμα ασφάλειας για μας. Γιατί ξέρετε ότι χιλιάδες ε, Ευρωπαίοι πολίτες ε, πήγαν στη Συρία για να πολεμήσουν ε, με το Ισλαμικό κράτος. Ξέρετε ότι πολλοί σκοτώθηκαν, αλλά πολλοί είναι ακόμη στην περιοχή. Και πολλοί από αυτούς τους τρομοκράτες θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν το χάος που έχει δημιουργηθεί για να επιστρέψουν στις χώρες μας. Τώρα, τα τελευταία χρόνια, έχουμε ελέγξει καλύτερα τα εξωτερικά μας σύνορα. Έχουμε περισσότερα στοιχεία για τους ε, ταξιδιώτες εντός και εκτός της Ένωσης. Αλλά έχουμε ακόμη την εντύπωση ότι η κατάσταση είναι ακόμη δυσχερής. Η Europol και τα κράτη-μέλη πρέπει να κάνουν πολύ περισσότερες προσπάθειες, διότι η ασφάλεια πρέπει να είναι η απόλυτη προτεραιότητά μας. Τέλος, η λεγόμενη σύμμαχός μας Τουρκία λέει ότι είναι δικό μας πρόβλημα αυτό η ασφάλεια. Ναι, αλλά κάθε χώρα πρέπει ακριβώς να ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Από κοινού μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της τρομοκρατίας. Ο κύριος Γκλούξμαν τώρα το λόγο για ένα λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, Έχουμε τα χαμόγελα των νικητών, τέδαμε χθε, στο πρόσωπο του Ερντογάν και του Πούτιν, αντικατοπτρίζουν πραγματικά τη δική μας τη δηλία. Και η Συρία αντιστοιχεί ουσιαστικά στην εγκατάλειψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγκαταλείψαμε τους Σύριους επαναστάτες στο όνομα της μάχης κατά του Άισις. Και στη συνέχεια εγκαταλείπουμε και τους καλύτερους συμμάχους μας στη μάχη αυτή κατά του Άισις, δηλαδή τις κουρδικές δυνάμεις. Σήμερα λοιπόν θα ρίξουμε όλη την ευθύνη στον Ντόναλτ Τραμπ και θα έχουμε απόλυτο δίκιο να το κάνουμε αυτό. Εμεί όμω, εμεί τι ακριβώ κάνουμε. Θα επιβάλλουμε κυρώσει, ναι, συμφωνώ και επαυξάνω, αλλά πότε. Πότε θα γίνει αυτό. Ήδη πυκνό σκοτάδι καλύπτει τη Συρία, ενώ εμεί βρισκόμαστε ακόμα στι αρχικέ δηλώσει. Πρέπει λοιπόν να αντλήσουμε τα διδάγματα τη αδυναμία μα. Και α το πούμε ξεκάθαρα, το ΝΑΤΟ δεν έχει πλέον νόημα, όχι επειδή δεν έχουμε αντιπάλου, αλλά γιατί δεν έχουμε πλέον έμπιστου συμμάχου. Α καταφέρουμε λοιπόν να δημιουργήσουμε μια αξιόπιστη ευρωπαϊκή άμυνα, να ελικιωθεί επιτέλου η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Βίκτορ Γκο έγραφε το ακόλουθο. Είναι ζωή μόνο αυτοί οι οποίοι μάχονται, αυτοί οι οποίοι έχουν ένα ανώτερο το οποίο γεμίζει την ψυχή τους. Οι φίλοι μας πεθαίνουν, σκοτώνονται και εμείς δεν είμαστε καν εν ζωή. Ο κύριος Γκέτα έχει το λόγο για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ας δούμε πώς έχουν τα πράγματα και στα κατονομάσουμε. Η ενδεχόμενη δημιουργία ενός Συριακού Κουρδιστάν ενδεχομένως να θεωρείται από την Άγκυρα ως μία απειλή για την εδαφική αικαιρεότητα της ίδιας της Τουρκίας. Αν δεν το συνειδητοποιήσουμε αυτό τότε ουσιαστικά θα μπορούσαμε να εξηγήσουμε καθόλου την παρουσία των κουρδικών δυνάμεων στη Συρία. Πρέπει λοιπόν να δούμε και την πτυχή αυτή. Και βέβαια πρέπει να συνειδητοποιήσουμε αυτή τη στιγμή ότι η στρατιωτική επέμβαση της Τουρκίας στη Συρία δεν μπορεί να γίνει αποδεικτή. Γιατί ουσιαστικά συμβάλλει περισσότερο στην οδύνη των δυνάμεων αυτών. Θα μείνει στην Συρία αυτή τη στιγμή ο Ερντογάν και θα αφήσει πίσω του ουσιαστικά μίσος και διάθεση για εκδίκηση Κατά αυτόν τον τρόπο, κύριε Ερντογάν, ενισχύεται το ΤΑΕΣ, το Ισλαμικό κράτος και ουσιαστικά δημιουργείται περισσότερες αντιπαραθέσεις δημιουργώντας μια πυρηταποθήκη στη Μέση Ανατολή. Πραγματικά δεν υπάρχει κανένας λόγος που να αιτιολογεί την πράξη αυτή του κύριου Ερντογάν. Κύριε ένα λεπτό. Αγαπητοί συνάδελφοι, μια σοβαρή ανθρωπιστική κρίση εκτελήσεται ταχεία στην ε, Ανατολική Συρία, ο Ερτογάν δεν μπορεί να αντέξει την δημοκρατική κοινωνία στην περιοχή και έχει δράσει βία. Βλέπουμε ε, πάνω από 200.000 ανθρώπους που αναγκάστηκαν να εκτοπιστούν, μεταξύ αυτών 70.000 παιδιά. Ακούσαμε από άλλους ομιλητές ε, τους λόγους για τους οποίους πρέπει να προστατέψουμε αυτά τα παιδιά και τους Κούρδους που δικαίως ζουν εκεί. Ε, δεν θα χαθεί μόνο η ζωή τους ή το σπίτι τους αν συνεχίσει η εισβολή. Ε, των Τούρκων. Ε, οι ακαδημαϊκοί, οι διαλυστές ε, σε όλο τον κόσμο έχουν θαυμάσει την περιοχή εκεί, την ύπαρξη των γυναικών που ζουν εκεί ειρηνικά με την γη τους. Θα πρέπει λοιπόν να πατάξουμε τον απολυταρχισμό και την στρατικοποίηση. Θα πρέπει να βοηθήσουμε τους γείτονες να μην ζουν υπό τις ίδιες απειλές. Είναι οι κυρώσεις που λειτουργούν οδηγούν σε αυτή την κατεύθυνση και τίποτα άλλο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για ένα λεπτό ο κύριος Τσόκα. Εντελώς τρελή, απαράδεκτη επέμβαση. Θα θυμάστε ότι στην προηγούμενη Ολομέλεια λέγαμε ότι ε, μας ζητούσαν να ξεκινήσουμε εκ νέου τις διαπραγματεύσεις για την ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή τη στιγμή, ενώ μας δίναν την προηγούμενη εβδομάδα σοκολάτες προκειμένου να καταφέρουμε εμείς να προχωρήσουμε με την ένταξη αυτή, αυτή τη στιγμή δεν δίνουν σοκολάτες, στέλνουν όμως όπλα, στέλνουν όλμους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτή τη στιγμή ως Ευρωπαϊκή Ένωση δεν καταφέραμε να διαχειριστούμε εμπορικού και άλλους πολέμους και χρηματοδοτούμε τρόπον την άφη τη στιγμή τον ίδιο τον στρατιωτικό πόλεμο που κάνει η Τουρκία. Ο Αντώνιο Μεγκαλίτσι είχε πει ότι ε, δεν, φτάνουν, δεν φτάνει το να τηρούμε ενό λεπτού σιγή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αν χρηματοδοτούμε έναν πόλεμο αυτή τη στιγμή, αν συμπράττουμε κι εμείς ε, κατά μάλλον υπέρ της Τουρκίας και κατά αυτών που έδωσαν μάχη κατά της τρομοκρατίας. Όσοι λάβανε αυτό το κουτί σοκολατάκια από την Τουρκία, ας το επιστρέψουν στην Τουρκία που τα χέρια της αυτή τη στιγμή είναι ματοβαμένα. Διακόπτεται. Σας παρακαλώ πολύ, καθίστε. Καθίστε, σας παρακαλώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Κοιτάξτε, βρισκόμαστε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είμαστε εδώ για να συζητάμε. Δεν βιοπραγούμε, δεν πετάμε αντικείμενα εδώ και εκεί. Είναι απαράδεκτη η συμπεριφορά σα. Δυστυχώ, συνάδελφοι, αυτά τα πράγματα πραγματικά γίνονται συνεχώς. Εδώ είναι κοινοβούλιο, εδώ συζητάμε. Δεν ε, χρειάζεται να φωνάζουμε, και να πετάμε πράγματα. Ελπίζω όλοι να συμφωνείτε. Με αυτό πραγματικά εξανίσταμε με αυτό που μόλις είδα. Είχατε το λόγο, παρακαλώ. Ακούστε με. Παρακαλώ, ακούστε με. Παρακαλώ, μπορείτε κύριε να ακούσετε ένα λεπτό. Γιατί καμιά φορά όταν ακούς μαθαίνεις. Η δικιά μου ε, δουλειά είναι να τηρώ την τάξη εδώ και αυτό που κάνατε ήταν κατά της τάξης ε, και ε, δεν σέβεται αυτό το κοινοβούλιο πραγματικά. Και καταχράστηκε το χρόνο των άλλων συναδέλφων. Συνεχίζουμε. Για ένα λεπτό, κύριος Λάμπακοφ. Κυρία Πρόεδρε. Διάβασα το σχέδιο ψηφίσματος ε, για «Η Τουρκία. Είναι ισχνά και ανεμικά. Δείχνουν την αδυναμία μας. Ε, λένε κάποια πράγματα με ακρίβεια, όμως ε, δυστυχώς αυτά τα μέτρα που προτείνουν δεν θα πετύχουν τίποτα. Προτείνω να παγώσουμε κάθε ευρωπαϊκή επένδυση στην οποία μπλέκονται τουρκικοί κυβερνητικά όργανα και θεσμοί. Νομίζω ότι αυτό πραγματικά θα πλήξει τον Ερτογάν γιατί ε, δεν γίνεται τα οικονομικά συμφέροντα πάντα να είναι πάνω από τις ανθρώπινες αξίες μας. Ε, ε, αυτά τα μέτρα θα είναι ένα μικρό τίμημα που θα πληρώσουμε για να σώσουμε τις ζωές χιλιάδων αθώων. Αν αυτά τα μέτρα πραγματικά τελικά αποδειχτούν επαρκή θα πρέπει να κάνουμε πλήρες εμπάρκο, να μην πουλάμε τα πινέζα. Ευχαριστώ για ένα λεπτό κύριος Μοργέλ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πραγματικά εισμάται είναι αυτές ε, οι ε, διαμαρτυρίες σήμερα. Έχουμε αφήσει στην άκρη τον ηρωικό αγώνα των Κούρδων και πραγματικά η λυπηρή αλήθεια είναι ότι εμείς ε, τους εγκαταλείψαμε, εμείς οι Ευρωπαίοι και δεν κάνουμε και πολλά πράγματα. Η επίθεση των Τούρκων εδώ και δύο εβδομάδες έγινε δυνατή ακριβώς λόγω της ε, ασυνέπειας ε, των Ηνωμένων Πολιτειών. Βλέπουμε τον Ερντογάν και τον Πούτιν τώρα να αποφασίζουν για τη μοίρα της περιοχής και να παγιώνουν είναι μεγαλύτερη ε, ηρωνία τον κύριο Μπασάρα Ελασάτ για τους Κούρδους ε, είναι δράμα, έχουν γίνει εργαλεία. Για τους Ευρωπαίους όμως είναι μεγάλη τροπή. Ήμασταν ανίκανοι να αντιδράσουμε σε μία μονομερή επίθεση και δεν μπορέσαμε να υπερασπιστούμε τους συμμάχους μας. Όμως πρέπει σήμερα να δούμε ακριβώς ε, και τι συμπεράσματα ε, βγάζουμε. Έχουμε ένα ΝΑΤΟ τελείως παράλογο που δεν έχει νόημα. Ε, η Ευρώπη είναι ανεξάρτητη, έχει την δύναμή της και εμείς καθόμαστε επιθύνια και υπακούμε στις παράλογες επιταγές των Αμερικανών. Δεν πρέπει να ρίχνουμε, να ρίχνουμε κροκοδίλια δάκρυα, απλώς να λαμβάνουμε σόφρονες αποφάσεις. Ένα λεπτό η κυρία Φεράρα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Η κυβέρνηση του Έρντογαν ξεπέρασε κάθε όριο ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι βυθίζεται σε μια αιματοχυσία. Η Μέση Ανατολή μια πραγματική τραγική ανθρωπιστική κρίση. Είναι οι Κούρδοι αυτοί που πληρώνουν το πιο υψηλό τίμημα. Θα πρέπει η διεθνή κοινότητα να δείχνει ευγνωμοσύνη για τη συμμετοχή του στην καταπολέμηση του ISIS. Αναφερόμαστε σε εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένου. αναφερόμαστε σε εκατοντάδες ε, μαχητέ του ISIS που έχουν βγει από τις φυλακές των Κούρδων. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή θα πρέπει να ασχοληθούμε λίγο περισσότερο με του βομβαρδισμού αμάχου πληθυσμού από μια χώρα η οποία παίρνει χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ελπίζει ότι ενταχθεί και μια μέρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν αρκούν όμω οι θεωρητικέ ε, κυρώσει μα. Θα πρέπει να προχωρήσουμε σε συγκεκριμένε κυρώσει. Η Ιταλία αποφάσισε να σταματήσει το εμπόριο όπλο προ την Τουρκία, αλλά κάτι ανάλογο θα πρέπει να κάνουν και οι υπόλοιπε χώρε Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει οποιαδήποτε χρηματοδότηση να σταματήσει και να σταματήσει επίση και η διαδικασία προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί ουσιαστικά η Τουρκία αυτή τη στιγμή στρέφεται κατά τη διαδικασία ειρήνευση και κατά των ίδιων των αρχών και των αξιών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Κυρία ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, είναι δύσκολο και έχει μεγάλη συγκινησιακή φόρτιση να συζητάμε αυτά που κάνει η Τουρκία και από τις δύο πλευρές των συνόρων της και αυτά τα οποία διαπράττει. Τα διαπράττει εδώ και πολύ καιρό. Να μην ξεχάσουμε ότι είναι χρόνια τώρα μετά τις φαγές που έγιναν στα Βαλκάνια. Να μην ξεχνάμε ότι η Τουρκία προσπαθεί να είναι όλο και πιο παρούσα ε, στην, περιοχή των Βαλκανίων. Δεν αρκεί να παγώσουμε τα περιουσιακά του στοιχεία. Πρέπει να δράσουμε πιο αποφασιστικά, να καταγγείλουμε τον Ερντογάν. Είναι ανήθικο αυτό που κάνει. Πρέπει να λογοδοτήσει ενώπιον του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Όπως όσοι διαπράττουν σφαγές και εθνοκάθαρση. Όπως έγινε στην Σρεμπρένιτσα ή στο Μπίχατς. Όλα αυτά, όλοι αυτοί που τα κάνουν αυτά τα πράγματα πρέπει να λογοδοτήσουν όπως είπα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Κάστε. ένα λεπτό. Ο πόλεμος ε, που κάνει το καθεστώς Ορντογάν στη Βόρεια Συρία είναι κατά του διεθνούς δικαίου και αποσταθεροποιεί την ευρύτερη περιοχή. Μέσω της απόσυρσης των Αμερικανικών στρατευμάτων βοηθούν οι Ηνωμένες στην Τουρκία. Τους άνοιξαν τον δρόμο. Η γεωπολιτική στρατηγική του Ερντοάν θέλει να καταργήσει τη Ροζάβα, την κουρδική αυτόνομη περιοχή και να διευρύνει την επικράτεια της Τουρκίας. Εδώ και χρόνια οι Κούρδοι καταπολεμούν επιτυχώς το Ισλαμικό κράτος. Αυτό είναι κάτι που συμβάλλει στην ασφάλεια και των δικών μας πολιτών. 11.000 ε, έχουν ε, πέσει στη μάχη κατά του Ισλαμικού κράτους. Εμείς τους οφείλουμε πολλά. Χαιρετώ ότι παρατείνεται το εμπάρκο όπλων, αλλά οι Κούρδοι, γυναίκες και άνδρες, πληρώνουν ένα πολύ βαρύ τίμημα. Δεν λαμβάνουμε όπως τα συμφέροντά τους. Η περιοχή απέχει μακριά από μια διαρκή ειρήνη. Τα πάνθρωπα σχέδια επανεκατάσταση του Ερντογάν πρέπει να καταδικαστούν. Πρέπει να δώσουμε μια προοπτική στους, Κόρδους, στους Κούρδους για μια αξιοπρεπή ζωή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η διεθνής κοινότητα πρέπει επιτέλους να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Ο κύριος ε, Τουντοράκα. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Όπως και οι συνάδελφοι καταδικάζω αποφασιστικά την ε, επιθετικότητα της Τουρκίας στη Βόρεια Συρία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δράσει. Ως εξή. Πρώτα απ' όλα σε ανθρωπιστικό επίπεδο. Υπάρχει ανθρωπιστική κρίση που ήδη είχε ιστορικά μεγάλες διαστάσεις και τώρα επεκτείνεται και οξύνεται είναι μια κρίση προσφύγων. Προστίθενται μερικές εκατοντάδες χιλιάδες στους ήδη υπάρχοντες πρόσφυγες. Επιπλέον, θα αποφεληθεί από το χάος του Ισλαμικό κράτος για να ανασυγκροτηθεί και θα απελευθερωθούν, αν δεν έχουν ήδη ελευθερωθεί, πολλοί από τους κρατούμενους του Ισλαμικού κράτους. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει πίεση από διπλωματικής πλευράς. Όχι μόνο γιατί ελέγχει στρατόπεδα προσφύγων. Πρέπει να το επιβάλλουμε να σέβεται το κράτος δικαίου. Μία Τουρκία που συνεργάζεται μόνο με τη Ρωσία πρέπει να λάβει σαφή μηνύματα από πλευρά Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να υπάρξει απαγόρευση πώληση όπλων. Πρέπει επίση να ενθαρρύνουμε την, την ε, τουρκική κοινωνία των πολιτών για να υπάρξει μια σταθεροποίηση και τη Συρία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ η κυρία Άουκεν για ένα λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, σε πολλές από τις χώρες μας έχουμε πολλούς Κούρδους που ζουν ε, για πολλά χρόνια ως πολίτες μας, ως κομμάτι της ε, πατρίδας μας, ως κομμάτι του εκλογικού μας σώματος. Νομίζω ότι έχουν έρθει πολύ κοντά μας και αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο Κουρδιστάν, γιατί ε, καταλαβαίνετε ότι έχουν στενούς δεσμούς με τις οικογένειές τους εκεί στην πατρίδα, είναι λυπηρό. Ε, δεν είναι ε, μόνο το γεγονός ότι το να υποφέρουν οι δικοί σου είναι χειρότερο από το να υποφέρουν οι άλλοι, αλλά και το γεγονός ότι εμείς πρέπει να λάβουμε υπόψη μας το γεγονός ότι χρειάζεται ειρήνη, όχι πόλεμος, όχι γενοκτονία. Δεν θέλουμε να πεθαίνουν τα παιδιά μας. Συνήθως λέμε ότι οι Κούρδοι έχουν για φίλους τους μόνο τα βουνά. Ας τους δείξουμε όμως ότι έχουν και άλλους φίλους. Ελπίζω σήμερα το ψήφισμα να συνεισφέρει σε αλλαγή πορείας, αλλαγή ρότας και να μην έχουμε μια κατάσταση σαν αυτή που φαίνεται ότι προκύπτει. Ευχαριστώ κύριος Ριβιέρ. Ε, κοιτάξτε, ε, πρέπει να υπάρχει μια ομόφωνη καταδίκη αυτών που κάνει η Τουρκία στο έδαφος ε, της Συρίας εδώ και πολλές μέρες. Σίγουρα πρέπει να καταδικάσουμε τον πόλεμο του Ερδογάν και τις φρικαλαιότητες που τον ε, ακολουθούν. Όμως θα πρέπει να χτυπήσουμε το κακό στη ρίζα του. Από το 2011 η Τουρκία αποσταθεροποιεί την ε, Αγγής Ανατολή και εμείς ε, κοιμόμαστε μπροστά στην εκβιασμό της Τουρκίας και του Πρόεδρου της. Τα δεχόμαστε όλα. Εσείς και ειδικά το ΕΛΚ λέτε ότι η Τουρκία ποτέ δεν θα μπει στην Ευρώπη. Εδώ στο Στρασβούργο συνεχώς όμως ψηφίζεται για περισσότερους πόρους στην Τουρκία. Δίνεται όλο και περισσότερους πόρους στον Ερδογάν. Ένα ε, σύνορο το οποίο είναι ελεύθερο εμπορίου δεν μπορείτε να το προστατεύσετε και πάτε όλο και πιο μακριά. Υπάρχει ένα διπλό παιχνίδι που στην ουσία αποκλείει οποιαδήποτε λύση σε αυτή τη σύραξη και μπαίνει και ο Πούτιν στο παιχνίδι. Πρέπει λοιπόν να σταματήσουμε να μένουμε εκεί άφωνοι και πρέπει να σταματήσουμε ε, τις ροές ε, που θα πρέπει των εκατομμυρίων που πρέπει τελικά να στεγνώσουν. Για ένα λεπτό ο κύριος Προκατσίνη έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Το δράμα το οποίο εκτιλήσεται για τους Κούρδους στη Συρία αποκάλυψε πολλές διαφορετικές ευρωπαϊκές υποκρισίες, μπορώ να πω. Η πρώτη είναι η εξή. Μολονότι χάναν τη ζωή του πάρα πολλοί Κούρδοι δίνοντα τη μάχη κατά του Άισι, εμεί καθόμασταν στον καναπέ και βλέπαμε τα γεγονότα στην τηλεόραση. Και τώρα ξαφνικά ανησυχούμε επειδή οι αλλοδαποί μαχητέ μπορεί να επιστρέψουν στην Ευρώπη, που είναι Ευρωπαίοι αυτό, μην το ξεχνάμε. Επίσης, ενώ όλα αυτά τα χρόνια η Τουρκία από κοσμικό καθεστώ, γινόταν σιγά σιγά Ισλαμικό Σουλτανάτο, 58 δισεκατομμύρια ευρώ έδωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση για να υποστηρίξει την προσχώρησή τη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τρίτη υποκρισία. Η απειλή του Ερντογάν ότι θα μα ρίξει τη βόμβα αυτή των προσφύγων ουσιαστικά έχει να κάνει με το ότι η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση επέτρεψε τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων τη να την αλάβει η Τουρκία. 6 δισεκατομμύρια ευρώ στήκησε αυτό. Και το λέω αυτό και προ τον Ευρωπαίο Επίτροπο. Καλέ κυρώσει κατά του Ερντογάν και τη κλίκα του, αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να σταματήσει τη διαδικασία προσχώρηση τη Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ο κ. Παπαδάκη, ένα λεπτό. Δεν πρόκειται για μονομερή στρατιωτική δράση όπως ισχυρίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά για την εισβολή στη Συρία του στρατηγικού της εταίρου, της Τουρκίας, κράτους μέλους του ΝΑΤΟ, με στόχο μερίδιο στον έλεγχο της περιοχής. Τόσο η Αμερικανοτουρκική Συμφωνία όσο και αυτή με τη ρωσία με όρους υπερελιστικής ειρήνης με το πιστόλι στον κρόταφο σηματοδοτούν νέο κύκλο παζαριών και ανταγωνισμών στις πλάτες των λαών τροφοδοτούν αβεβαιότητα για τους λαούς στο πλαίσιο στρατιωτικής κλιμάκωσης στην περιοχή είναι υποκριτικέ οι κυρώσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση τόσο για την εισβολή στη συρία όσο για τι παραβιάσει σε αιγαίο και κυπριακή αόζ ενώ οικονομικέ, εμπορικέ και άλλε σχέσει ισχυρών κρατών μελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση αναβαθμίζονται και ενισχύονται. ευρωπαϊκή ένωση ηπα νατο οι υπερελιστέ συνολικότερα δεν πιάνονται φίλοι όπω ισχυρίζονται η κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία και ο σύριζα στην ελλάδα. οι συμμαχίε του είναι σε βάρον των λαών αλληλεγγύη στον κούρδικο πληθυσμό και συνολικά στο συριακό λαό να τερματιστεί η επίθεση των τουρκικών στρατιωτικών δυνάμεων. η εξελίξη στη συρία είναι υπόθεση του λαού της. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Κόβατσεφ έχει το λόγο τώρα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τα όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στην βορειοανατολική Συρία δημιουργούν πάρα πολλές ανησυχίες και αποτελούν και μια προειδοποίηση για το τι συμβαίνει τελικά όταν δεν υπάρχει ισχυρή εξωτερική πολιτική και όταν δεν υπάρχει απαραίτητη ικανότητα ανάληψης δράσης στις γειτονικέ μας περιοχές. Είμαστε πάρα πολύ καλοί στο να κάνουμε δηλώσεις, αλλά τελικά όχι τόσο καλοί στο να λαμβάνουμε δράση, έτσι δεν είναι. Η Ρωσία, από την άλλη, φαίνεται ότι μπορεί και εκμεταλλεύεται πολύ καλά σας ζητώ συγγνώμη που σας διακόπτω. Να προσπαθήσουμε μία ακόμα φορά. Συγγνώμη. Σας ακούω αυτή τη στιγμή. Πολύ ωραία. Κυρία Πρόεδρε, σας έλεγα ότι η στρατιωτική επιχείρηση της ε, Τουρκίας ουσιαστικά θέτει να αμφιβόλο την περιφερειακή ασφάλεια καθώς επίσης και την καταπολέμηση του Ντάεσ. Νομίζω ότι θα πρέπει να καταφέρουμε να επέμβουμε με τρόπο πολιτικό και διπλωματικό συνεργαζόμενοι με τους συμμάχους του ΝΑΤΟ από το να επιρρύπτουμε μερό την ευθύνη εδώ και εκεί. Βλέπετε ότι αυτή η εκεχηρία, προσωρινή εκεχηρία δεν σταμάτησε την ανθρώπινη οδύνη όλων αυτών των ανθρώπων που κατοικούν στην περιοχή, είτε μας αρέσει είτε όχι. Η Τουρκία αποτελεί εταίρο μας. Είναι λοιπόν προς το δικό μας το συμφέρον να κρατήσουμε την Τουρκία στην ευρωπαϊκή της προοπτική, αρκεί βέβαια να τηρεί τις δεσμεύσεις της. Και βέβαια οι όμορες της, χωρι... της Τουρκίας χώρες χρειάζονται και την αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως η Ελλάδα και η Βουλγαρία. Ο κύριος Σίντερ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η στρατιωτική επέμβαση της Τουρκίας ε, είναι κατά του διεθνούς δικαίου πρώτον και εσωτερικά κινητοποιημένη γιατί ο Ερδογάν έχει χάσει πολλές εκλογές τελευταία. Οι συνέπειες είναι μασική φυγή πολιτών, χριστιανών, σύρων, αρμένιων. Ε, πάνω από 200.000 άνθρωποι έχουν βγει στο δρόμο, 70.000 παιδιά. Υπάρχει κίνδυνο στο Ισλαμικό Ισλαμικό κράτος να ενισχυθεί και πάλι και ε, ε, να πω ότι ε, το YPG δεν είναι τρομοκράτες, είναι αυτοί που απελευθέρωσαν την περιοχή από το Ισλαμικό κράτος. Χρειαζόμαστε λοιπόν εκεχηρία, μια διπλωματική επέμβαση, μια αποστρατικοποιημένη ζώνη, η ανθρωπιστική βοήθεια, εμπάργκο όπλων, κυρώσεις κατά της Τουρκίας και μια συζήτηση για το αν θα πρέπει να συνεχίσουν οι διεξιακές διαπραγματεύσεις και μια αλληλεγγύη με την αυτοδιοικούμενη περιοχή των Κούρδων στη Ροζάβα. Για ένα λεπτό, ο κύριος Πέλιον. Ε, Ευχαριστώ. Η απόσυρση των, των στρατευμάτων των ΗΠΑ είναι η μεγαλύτερη προδοσία όλων των καιρών. Πριν από ένα χρόνο ο Τραμπ είπε στους Κούρδους ότι αυτοί ε, μάχονται, είναι εξαιρετικοί άνθρωποι, δεν το ξεχνάμε και εγώ δεν το ξεχνώ. Σήμερα είναι η ε, ανόητοι οι Τούρκοι, ε, οι χρήσιμοι ανόητοι στην εξυπηρέτηση των Αμερικανών. Είναι πραγματικά ανεύθυνη αυτή η στάση. Η Τουρκία ε, πραγματικά μιλάει για δύσκολες αποφάσεις, αλλά καλά θα έκανε να κοιτάξει το δικό της έδαφος ε, και να δώσει περισσότερο χώρο στην αντιπολίτευση που υποστηρίζουν τους ε, Κούρδους και στους δημοσιογράφους που υποστηρίζουν τα δικαιώματά τους και να μην τους λέει οι τρομοκράτες. Χρειαζόμαστε μια πολιτική λύση που θα επιτρέψει την επιστροφή των εκτοπισμένων ε, και θα μειώσει το στρατηγικό χώρο που δίνεται και παραχωρείται στην Ρωσία, τον Ασάτ και το Ιράν. Ευχαριστούμε για ένα λεπτό κυρία Τσεκάρντι έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πριν από 100 χρόνια οι Αρμένοι αποτέλεσαν το ίστατο θύμα της Τουρκίας και αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι ανάλογη είναι η στάση των Τούρκων απέναντι στους Κούρδους και βλέπουμε ότι χύνεται ακόμα αίμα αθώων, όπως για παράδειγμα τη Καλέβη, η οποία ήταν Κούρδος πολιτικός που μιλούσε υπέρ των δικαιωμάτων των γυναικών και που εκτελέστηκε ουσιαστικά από τους φιλοϊσλαμιστές συμμάχους της Τουρκίας. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι όλο και περισσότερο φτάνουν οι μαχητέ του ISIS στι πόρτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση εξαιτία τη κατάσταση στη βρονταλική Συρία και τη εισβολή τη Τουρκία. Και ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή μα απειλεί ακόμα περισσότερο, μολονότι έχει λάβει από εμά 6 δισεκατομμύρια ευρώ. Μα απειλεί ότι θα ανοίξει τι πύλε και θα μα κατακλείσει με, με πρόσφυγε. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε, η Ρωσία γίνονται οι βασικοί πρωταγωνιστέ, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση για μία ακόμα φορά σιωπεί και αποτελεί έναν απομακρυσμένο παρατηρητή. Είναι πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι ανάλογη απαθή είναι και η Φεντερίκα Μογκερίνη και Ντρέπομαι πραγματικά που είναι από την ίδια χώρα με μένα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε αυτή τη στιγμή ότι όσο χρηματοδοτούμε την Τουρκία γινόμαστε συνένοχή τη. Όχι, ποτέ Τουρκία στην Ευρώπη. Τελεί και παύλα. κύριο Ευχαριστώ πολύ. Θεωρώ ότι είναι άθλιος ο τρόπος με τον οποίο κάνουμε εδώ κοινικές ομιλίες ενώ γίνονται αυτά τα άθλια στη Συρία. Πραγματικά, σκεφτείτε τι λέτε. Ο κουρδικό λαός προδόθηκε. Μας βοήθησε κατά του Ισλαμικού κράτους και τώρα τους ε, εγκαταλείπουμε. Και οι Αμερικανοί με την απόσυρση των δυνάμεών τους επιτρέπουν την εισβολή τη Τουρκία. Όλοι ήξεραν ότι η Τουρκία πρόκειται να εισβάλλει μόλι θα αποσύρονταν οι Αμερικανοί. Ε, τα δεινά των ε, κατοίκων της Συρίας πρέπει να σταματήσουν οι αξίες μας και το πώς αποδίδουμε το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης μας ε, υποβάλλουν να τονίσουμε ότι όχι δεν είναι ε, επέμβαση ειρήνης αυτή, είναι έγκλημα πολέμου. Οι, δικτατόρ, οι δικτάτορες δεν πρέπει να έχουν θέση στις σχέσεις μας. Πρέπει να το καταστήσουμε σαφές για άτομα τα οποία δεν επιτρέπουν την ελευθερία του τύπου, της θρησκείας, ε, της πολιτικής σκέψης, όπου έχουμε τόσο όλο και περισσότερους ε, πολιτικούς ε, κρατουμένους στις φυλακές δεν πρέπει να έχουν σχέση μαζί μας. Η διπλωματία είναι αναγκαία αλλά χρειάζονται και κυρώσεις σε κάθε επίπεδο. Πρέπει να εκφραστεί σαφώς η Ένωση. Χρειάζονται κυρώσεις, όχι μόνο διπλωματία. Δεν το διαπιστώνω αυτό. Είναι σημαντικό η Ευρώπη να μιλήσει με ενιαία φωνή. Διακόπτε το μιλήτες. Ο κύριος Γκιόγκιωση, ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πολλοί αναφέρθηκαν στην έλλειψη ενότητας στην Ένωση. Την αποτυχία μας να υπάρξει έστω μια κοινή δήλωση που να καταδικάζει την τουρκική επιθετικότητα. Η Ουγγαρία όμως άσκησε βέτο σε αυτή την κοινή δήλωση ως ε, Ούγγρος ζητώ συγγνώμη και καθιστώ σαφές ότι όταν μιλάω Βίκτορ Όρμπαν από πλευρά των Ούγγρων δεν μπορείτε να δέχεστε αυτά που λέει. Σας διαβεβαιώ ότι δεν είναι προ το συμφέρον ούτε των Ούγγρων, ούτε τη χώρα μου, να στηρίζουμε αυτές τις επιθέσει οπουδήποτε και αν συμβαίνουν. Όχι, δεν είναι προ το συμφέρον των Ούγγρων και αυτή η στρατιωτική επέμβαση της Τουρκίας ναι, μεν καταλαβαίνουμε τι ανησυχίε ασφάλεια τη Τουρκία, αλλά δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστεί με στρατιωτικό τρόπο αυτό το πρόβλημα, μόνο με πολιτικά και διπλωματικά μέσα. Αυτή η επίθεση αποσταθεροποιεί περαιτέρω τη Συρία, παρεμποδίζει την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και επιδεινώνει την μεταναστευτική κρίση. Πολλοί διαρωτώνται τι έχει κάνει η Ένωση. Εμείς είμαστε στο περιθώριο. Είμαστε παρατηρητές ενώ η γειτονία μας αποσταθεροποιείται στην ε, Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική. Η Ευρώπη πρέπει να επανέλθει στη δράση. Πρέπει να παίξουμε μεγαλύτερο ρόλο πριν άλλε κυρίαρχε δυνάμει. Διακόπτε το μιλητή. Ευχαριστώ πολύ, λέει πρόεδρο. Ο κύριο Μπελαμή, ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ. Η αγανάκτηση βεβαίω είναι ευρέω διαδεδομένη, αλλά δεν αρκεί. Αυτό που διακυβεύεται είναι η ειρήνη στη Μέση Ανατολή, αλλά και η δική μα ασφάλεια. Γιατί ο κύριο Ερντοάν είναι ο πρώτο σύμμαχο του Ισλαμικού κράτου με αυτά που κάνει. Η επίθεση που κάνει θα έχει επιπτώσει στην επικράτειά μας. Και όμως είμαστε ανίκανοι να αντιδράσουμε. Ας το αναγνωρίσουμε. Αυτή η σιωπή είναι απόδειξη της ανικανότητάς μας. Δεν έχουμε τις στρατηγικές δυνατότητες άμυνας. Δημιουργήσαμε μια αγορά αντί να βασιζόμαστε σε αρχές του κοινού μας πολιτισμού. Και γιατί είμαστε ανίκανοι να καθορίσουμε ελεύθερα την μεταναστευτική μας πολιτική. Γίνονται εκβιασμοί από πλευράς Ερντοάν για το θέμα της μετανάστευσης. Και αυτό αποδεικνύει την ανικανότητά μα να ελέγξουμε τα εξωτερικά μα σύνορα. Άρα είμαστε ανίκανοι να συμβάλλουμε και στι παγκόσμιε ισορροπίε. Πρέπει επιγόντω να έχουμε τα μέσα για να δράσουμε. Δεν μπορούμε να είμαστε θεατέ παγιδευμένοι σε αυτή την ανικανότητα. Πρέπει να σταματήσει η δηλία μα. Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να υποχρέσουμε την Τουρκία να διαπραγματευτεί. Πρέπει να σταματήσουν τάχιστα οι πόροι που παρέχονται στη χώρα αυτή. Δεν έχουν να κάνουν με ένα πρόγραμμα ένταξη τη χώρα. Ευχαριστώ πολύ. Ένα λεπτό ο κύριος Παπαδάκης. Η Τουρκία προβαίνει σε εθνοκάθαρση με στόχο την εξαφάνιση του κουρδικού στοιχείου από την περιοχή αξιοποιώντας το χώρο που έδωσαν οι Αμερικανοί με την αποχώρησή τους. Όλοι είναι παρόντες στην περιοχή με μεγάλο απόντα την Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία στο τέλος της ημέρας εκτός από τα θύματα των τουρκικών θηριωδιών είναι αυτή η οποία πληρώνει το λογαριασμό χωρίς να μπορεί να πάρει την όποια πρωτοβουλία για να σταματήσει η τουρκική εισβολή. προφανώς οι οικονομικές συναλλαγές χωρών της ευρώπης έχουν μεγαλύτερη σημασία από την προστασία του κουρδικού λαού που είναι αυτός που πολέμησε τον ντάεσ. δεν είναι δυνατό ολόκληρη η ευρωπαϊκή ένωση να συνεχίζει να παραμένει όμηρος στους εκβιασμούς ερντογάν. Ε, Για ένα λεπτό τώρα κυρία Ρίση έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Οι Κούρδοι μαχητές, Άραβες, Χριστιανοί, Τουρκμένοι έδωσαν μια μάχη στο όνομα της ανθρωπότητος. Η δική μας η ανθρωπιά που βρίσκεται ο Βεριβάν Ναντουιζέλ το λέει αυτό, μια Βελγίδα μάλλον πολίτης, Κούρδος, Ευρωπαία πολίτης, που απευθύνεται σε εμά σήμερα το πρωί και όλοι μας σήμερα είμαστε Κούρδοι απέναντι στην παράνομη αυτή στρατιωτική επέμβαση της Τουρκίας στην βροντολική Συρία. Βλέπουμε τις αποφάσεις αυτή τη στιγμή που λάβανε Αμερικάνοι, Τούρκοι και Ρώσοι. Και βλέπουμε πώ οι αποφάσει αυτές τρέφονται κατά των ανθρώπων αυτών που δώσανε μία μάχη για τη δική μας την ελευθερία. Και νομίζω ότι είναι τραγική ηρωνία αυτή τη στιγμή ότι ουσιαστικά εμείς ενισχύουμε τους ίδιους τους εχθρούς της δημοκρατίας. Το να θεωρούμε ότι νομοποιείται πλέον η δράση του Μπασάρα Λασάτ αποτελεί τραγική ηρωνία. Πού βρίσκεται σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο οι Ευρωπαίοι ηγέτες δεν έχουν εγκαταστήσει ένα ευρωπαϊκό εμπάργο πώληση όπλων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε αυτή τη στιγμή να παγώσουμε οποιαδήποτε χρηματοδότηση προς την Τουρκία, χωρίς να θέτουμε όμως σε καμία περίπτωση εν κινδύνο τον άμαχο πληθυσμό που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη Συρία. Ο κύριος Κοφώτη έχει το λόγο για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή απειλεί την Ευρώπη ότι θα αποστείλει εκατομμύρια πρόσφυγες προς την Ήπειρό μας. Το σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αποτύχει. Έχουμε δώσει τον έλεγχο των εξωτερικών μας συνόρων, τον έχουμε παραχωρήσει στον Ερντογάν. Παράλληλα βλέπουμε ότι δίδονται και όλα περισσότερο χρήματα των Ευρωπαίων φορολογουμένων προς τα ταμεία του Ερντογάν. Έχουμε αποτύχει τελικά να προστατεύσουμε παράλληλα και τα εξωτερικά μας σύνορα, τα οποία είναι διαπερατά. Ενώ απειλούμεθα ουσιαστικά με τις ίδιες απειλητικές καταστάσεις που είχαμε και το 2015, όταν θα θυμάστε τότε η Ευρώπη έπρεπε να αντιμετωπίσει ένα ισχυρότατο προσφυγικό κύμα. Πολύ φοβάμαι ότι καθώς πλησιάζουν τα Χριστούγεννα θα δούμε όλο και περισσότερους τρομοκράτες του ISIS οι οποίοι θα επιστρέφουν στις ευρωπαϊκές πόλεις, στις χριστουγεννιάτικες μας αγορές. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να σταματήσει αυτή η συνεχής ροή ευρωπαϊκών κονδυλίων προς το καθεστώς Τερντογάν ο οποίο πραγματικά θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνε του. Η κυρία Ντούρι Νικολσόνοβα έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κοιτάξτε, εγώ ήμουν πάντα ε, υπέρ του εγχειρήματο Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά τώρα λυπάμαι για τη δηλία μα. Πετάξαμε του Κούρδου ε, στα σκουπίδια. Ο Τραμπ ε, απέσυρε τι δυνάμει του αλλά κοιτάξτε, εμεί είμαστε πιο κοντά στη Μέση Ανατολή από ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε. Πού είναι οι δικέ μα ε, στρατιωτικέ μονάδε. Η πολιτική μα ε, εξωτερικών και ασφαλεία είναι αδύναμη. Είμαστε κομπάρσι. Είμαστε θεατέ, ούτε καν κομπάρσι. Δεν κάνουμε τίποτα. Οι μόνοι που παίζουν ρόλο συζητούν με τον Πούτιν, όχι με εμά. Εμά μα αφήνουν να παρατηρούμε τον Ερντοάν να εισβάλλει και να μας επιβάλλει την πολιτική του. Οι χώρες του Βίσεγκραντ το τόνισαν εδώ και νωρίτερα. Τα προβλήματα πρέπει να λύνονται εκεί που προκύπτουν. Τι περιμένουμε λοιπόν. Θα πρέπει να αντρέπομαστε για αυτά που κάνουμε. Όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτή τη δηλία μας στο Κούρτισαν. Ευχαριστώ πολύ. Φίλιπς, ε, ένα λεπτό. Το Ηνωμένο Βασίλειο επιτέλους σταμάτησε τι εξαγωγέ όπλων στην Τουρκία. Αλλά είναι πολύ λίγο και πολύ αργά αυτό. Θέλουμε τώρα και οικονομικέ κυρώσει. Αλλά τι μπορούμε να κάνουμε, ενώ συνεχίζουμε να πληρώνουμε σε αυτό το αδίστακτο κράτο για να χρηματοδοτεί ε, τον επεκτατισμό του. Δεκάδε χιλιάδε Κούρδοι ήταν στο πλευρό μα για να προστατεύσουν από την κτηνότητα τρομοκρατία και χιλιάδε έδωσαν τη ζωή του. Θα πρέπει να αμυφθούν. Αντί γι' αυτό η Ένωση δεν κάνει τίποτα ενώ ο Ερντοάν χρησιμοποιεί τη δωροδοκία των, της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να δολοφονήσει τους πολίτες, τον άμαχο πληθυσμό. Τι αξία έχει η ζωή ενός Κούρδου, τα 1500 που δίνουμε στην Τουρκία ή τι 160.000 εκατομμύρια Κούρδων που έχουν μετατοπιστεί. Αν τα συγκρίνουμε όλα αυτά, κοστίζει ένα λεπτό η ζωή ενός Κούρδου. Αυτό είναι μια ιστορική προδοσία η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ηθικά πτωχευμένη. Είναι ντροπή αυτά που κάνετε. Όλοι συμφωνούμε. Πρέπει λοιπόν να κάνει κάτι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί αλλιώ τι έννοια έχει να βρισκόμαστε εδώ μέσα. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ραντζέο. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Καταρχάς, Πρέπει να σας πω ότι ε, παρακολούθησα πολύ προσεκτικά τις ε, παρεμβάσεις των συναδέλφων, τις παρεμβάσεις που γίνανε σήμερα, οι οποίες σχεδόν όλες ε, καταδικάζουν απερίφραστα την στρατιωτική εισβολή της Τουρκίας στη βορνοτολική Συρία, που έχει οδηγήσει στον εκτοπισμό πάρα πολλών Κούρδων, που έχει δημιουργήσει με ένα καθεστώς αιματοχυσίας και πάρα πολλές παραβιάσεις ε, του ανθρωπιστικού και διεθνούς δικαίου. Και βέβαια πρέπει να πούμε ότι ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδίως το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα πρέπει να λάβει πιο δραστικά μέτρα κατά της επιθετικής αυτή τάσης του Ερντογάν. Εγώ ανησυχώ όμως πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Γιατί αρχίζω και θυμάμαι κάποια πράγματα τα οποία συνέβησαν στο παρελθόν. Η συμφωνία αυτή Ερντογάν-Πούτιν ξυπνά κάποιες ιδεχθείς ιστορικές μνήμες. Δεν μπορούμε να αφήσουμε το μέλλον της Συρίας ανάμεσα σε δύο δικτάτορες, τον Ερντογάν και τον Πούτιν. Έχουμε δει τέτοια ανάλογα παραδείγματα στο παρελθόν και γνωρίζουμε ότι τα αποτελέσματα ήταν τραγικά για όλους τους εμπλεκόμενους πληθυσμούς. Σας ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε ο κύριος Πιζαπία τώρα έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ζουν όλοι με αγωνία και με θυμό, με οργή, την στρατιωτική αυτή δράση της Τουρκίας κατά της Συρίας. Πρόκειται πραγματικά για ένα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, για μια πράξη πολέμου. Προδώσαμε ως διεθνής κοινότητα τους Κούρδους. Γυρίσαμε την πλάτη στους Κούρδους. Η συμφωνία Έρντογαν-Πούτιν αποτελεί ένα ακόμα βήμα υποτίθεται προς τη δημοκρατία και προς την ελευθερία. Πρέπει να το σταματήσουμε αυτό. Δεν φτάνει μόνο να αποκλείσουμε τις εξαγωγές όπλων. Χρειάζεται πραγματικά περισσότερο θάρρος. Και έλεγε και ο Νερούδα ότι πραγματικά θα πρέπει να μπορεί κανείς να έχει θάρρος, αλλά να μπορεί να αποδοκιμάζει και όλα στα κακό σκήμενα. Θεωρώ λοιπόν ότι το ψήφισμα το οποίο θα εγκρίνουμε σήμερα είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα, αλλά είναι θεωρητικό. Θα πρέπει να περάσουμε στις πράξεις. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε μια ζώνη απαγόρευσης πτήσεων. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε τους απαραίτητους ανθρωπιστικούς διαδρόμους. Θα πρέπει να επιβάλλουμε στοχευμένες οικονομικές κυρώσεις κατά της Τουρκίας. Αν δεν το κάνουμε τώρα, πότε θα το πράξουμε. Ο κύριος Χουκ για ένα λεπτό. Η επίθεση της Τουρκίας εναντίον των Κούρδων στη Βόρεια Συρία είναι πραγματικά καταστρεπτική. Έχουμε ιατροφαρμακευτική σε εγκαταστάσεις, την πρόσβαση στο καθαρό νερό, όλα αυτά καταστρέφονται. Αυτά επιτρέπουν στον ISIS να αναζωπηρωθεί και επιπλέον να αποσταθεροποιήσει την περιοχή. Κάποια κρατημέλη άμεσα πουλούν ε, όπλα ε, στην Τουρκία. Οι ευρωβουλευτές ε, των Ελεύθερων Δημοκρατών έχουν γράψει ήδη και ζητούν να σταματήσει αυτή η γενοκτονία. Έχουμε μιλήσει για τις νέες άδειες για πώληση όπλων, αλλά γίνεται με αυτές που ήδη έχουν δοθεί. Έχουμε κάνει μόνο το μισό δρόμο και αυτό είναι απαράδεκτο. Ο Τραμπ υποστηρίζει αυτές τις δράσεις. Εμείς θέλουμε να έχουμε μια ισχυρή, ε, αποτελεσματική Ευρώπη. Αν θέλουμε να είμαστε ενάντια αυτών που διαπράπτουν τα εγκλήματα, πρέπει να τους εμποδίζουμε να τραβούν τη σκανδάλη. Έχει έρθει λοιπόν ο καιρός να σταματήσουμε την υποψηφιότητα της Τουρκίας ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κυρία Λίτση για ένα λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, δεν είναι μόνο οι Κούρδοι οι οποίοι κινδυνεύουν και προ οποίου πρέπει να δείξουμε αλληλεγγύη. Η τουρκική αυτή επίθεση ενδεχομένω να οδηγήσει στην εξάλληψη τη χριστιανική κοινότητα που βρίσκεται εδώ και δύο χιλιετίε στη Συρία και αποτελεί ένα απόσπαστο τμήμα του κοινωνικού τη ιστού. Η υπεράσπιση των χριστιανών εντό και εκτό του χώρου Σέγγεν αποτελεί υποχρέωση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορούμε αυτόν το αμελήσουμε. Η Ευρώπη θα πρέπει να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο υπερασπιζόμενη την ειρήνη στη